So uh, Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Θέλω πρώτα απ' όλα να σας επισημάνω ότι τα συνοπτικά πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης έχουν ήδη διανεμηθεί και να ρωτήσω εάν υπάρχουν παρατηρήσεις Διαφορετικά θα θεωρήσω ότι τα συνοπτικά πρακτικά έχουν εγκριθεί. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Όμπερμαϊερ ε, που ε, έχει ζητήσει να θέσει ένα διαδικαστικό ζήτημα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω ένα σημαντικό θέμα επί της διαδικασίας και παρακαλώ να μου δοθεί απάντηση. Έχω μεγάλη κατανόηση και συμπάθεια για πολλούς ακτιβιστές που είναι αντίθετοι με την Συμφωνία Άκτα. Θα ήθελα να μάθω εάν πρόκειται να γίνεται δεκτό για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως να γίνονται δράσεις διανομής φυλαδίων κλπ. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό να ξεκαθαριστεί, να έχουμε μια πληροφορία. Εάν δηλαδή και στο μέλλον θα πρέπει να τηρούμε κάποια ε, στάση. Πώς, τι στάση θα κρατούμε όταν υπάρχουν μάλιστα και ομάδες επισκεπτών. Θα ήθελα μια απάντηση, ενώ σήμερα τουλάχιστον να μου διαβιβαστεί αργότερα κύριε Ομπερμάγερ. Συγκρατούμε την παρατήρησή σας. Να σα επισημάνω καταρχήν ως πρώτη αντίδραση ότι σε ό,τι αφορά τη διανομή φυλαδίων εκτό της αιθούσης δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Δεν εντοπίσαμε ε, να έχει δημιουργηθεί κάποιο ζήτημα ε, ενάντια στου κανονισμούς ε, σε ό,τι αφορά τη διανομή υλικού εντό της αιθούσης. Άρα καταρχήν το Προεδρείο εκτιμά ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αλλά οπωσδήποτε σας διαβεβαιώνω ότι θα το διερευνήσουμε περαιτέρω. Ε, Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η σύσταση του κυρίου Μάρτιν Εμπορική Συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης, απομίμησης